Αραβίας. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Uh, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, α, να αφήσω την κυρία Επίτροπο να καταλάβει τη θέση της. Ναι, σας Δείξω λίγη ευγένεια. Uh, <clears throat> Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόκειται για ένα χειρισμό, ή μάλλον μια χειρονομία ε, συμβολική από αμυγός οικονομικής άποψης, αλλά είναι πολύ μεγάλης πολιτική σημασία σε μια κρίσιμη ιστορική ε, στιγμή για τη Μολδαβία και την ολόκληρη γειτονία μας. Για τη Μολδαβία είναι μια ανάσα ε, νέου αέρα σε, μια, σε ένα πολύ σημαντικό τομέα την καλλιέργεια οποροκυπευτικών. Εκτός από τα μήλα όμως και τα άλλα φυτά που θα σας αναφέρω στη συνέχεια, ε, αυτό επιδεικνύει αλληλεγγύη σε πολύ χαλεπούς καιρούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μολδαβία στις 27 Ιουνίου υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης. Η Μολδαβική Βουλή στις 2 Ιουλίου αμέσω μετά έσπευσε να την κυρώσει και όλος τυχαίω, ε, ε, αμέσω μετά η Ρωσία επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής γεωργικών προϊόντων από τη Μολδαβία και στις 2 Αυγούστου απαγόρευση απαγόρευσε και από την την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Αγωγή τροφίμων στα πλαίσια ε, της Ουκρανικής κρίσης που βεβαίως ε, συνδέεται με το θέμα της Ανατολικής Γειτονίας. Πού ε, είναι η αιτία του κακού. Εσφαλμένα θεωρεί η Ρωσία ότι είναι θύμα κάποιας γεωπολιτικής συνωμοσίας της Δύσης. Εδώ πρόκειται για το 19ο αιώνα που πολεμάει τον 21ο αιώνα. Ε, ε, η προπαγάνδα, τα ψέματα, η εσωτερική διάβρωση και τα μήλα ξαφνικά έγιναν το μήλο της έρηδος γενικότερα. Και οι μολδαβικές αρχές ε, αναζήτησαν επίγουσα υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί ο αντίκτυπος της απαγόρευσης για τα πιο σημαντικά προϊόντα που είναι τα επιτραπέζια σταφύλια, τα μήλα και τα δαμάσκηνα. Ε, ε, ε, συμφώνησε το Συμβούλιο και ελπίζω το Κοινοβούλιο να δώσει επίσης τις ευλογίες του αυτή την εβδομάδα. Η απαγόρευση πλήττει δραματικά την οικονομία. Η γεωργία είναι περίπου 40% του ΑΕΠ τους και τα οποροκυπευτικά και μόνο έχουν 250.000 εργαζόμενους που συνιστά το 10% του ενεργού πολιτισμού της Μολδαβίας που προφανώς ζουν στην Ήπεθρο και καλλιεργούν μικρομεσαίες ε, εκτάσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις είναι. Ε, οι αυτόνομες λοιπόν εμπορικές προτιμήσεις τι είναι. Είναι ένα μέσο που έχουμε ε, τη δυνατότητα ένας εμπορικός εταίρος να παρέχει κάποιες επαναχωρήσεις σε μια χώρα για να υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή και την οικονομία χωρίς ανταλλάγματα. Το 2008 ήδη αρχίσαμε το εφαρμόζουμε αυτό απέναντι στη Μολδαβία με τον κανονισμό που τώρα τροπολογούμε. Ε, προτείνονται τώρα τρία νέε προ 40.000 μήλα, 20.000 ε, ε, τόνοι επιτραπέζια σταφύλια και 20.000 τόνοι δαμάσκηνα. Οι προστώσεις αυτέ είναι προσωρινέ και αφορούν το παράρτημα 3 και είναι σχετικά περιορισμένα σε σχέση με την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 0,4% της δικής μας παραγωγής είναι τα μήλα και είναι πολύ διαφορετική και η κλάδη της αγοράς που απευθύνονται. Και ιδιαίτερα λόγω της ε, κουλτούρας και της γεωγραφικής εγκύτητας με τη Ρουμανία, ε, περισσότερες ε, ποσότητες αυτές και των τριών προϊόντων εύκολα απορροφώνται από την ρουμανική αγορά. Για τα μήλα φέτος η Ρουμανία έχει μείωση στην παραγωγή 22% και σε σχέση με την ποσόστοση αυτή που μιλούμε είναι μόνο το 8% της ρουμανικής παραγωγής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα απορροφηθεί. Να πω και δύο λόγια τώρα στα ρουμανικά. Ε, έλεγα λοιπόν ότι ε, οι, οι μολδαβικές αρχές ε, θα προσπαθήσουν και θα επιτύχουν πιστεύω να ε, μετατρέψουν αυτή την υπόθεση σε μια δική τους νίκη. Ε, κάνω έκκληση προς τις ρουμανικές αρμόδιες αρχές να υποφεληθούν από το εμπόριο με τη Μολδαβία και βεβαίως ε, τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Ευχαριστώ κύριε Μόησα. Η Επίτροπος κυρία Μάλστρομ έχει το λόγο και σας καλωσορίζω γιατί για πρώτη φορά ε, προεδρεύω εγώ και έχω την ευκαιρία σας δίνω το λόγο σε επίτροπο. Κυρίες και κύριοι αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, η προσοχή των μέσων ενημέρωσης αφορά κυρίως την Ουκρανία. Υπάρχει όμως και άλλη μια γειτονική χώρα στην περιοχή, η Δημοκρατία της Μολδαβίας που αντιμετωπίζει τις πολιτικές συνέπειες της επιλογής που έκανε να υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας ξέρει ότι η οικονομική της ανάκαμψη ε, και ανάπτυξη θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι κάτι το οποίο δεν το έκανε η Μολδαβία εναντίον κάποιου άλλου, αλλά τώρα τα προϊόντα που πήγαιναν στη Ρωσία δεν μπορούν πια να εξαρθούν και οι παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις και με τις υπόλοιπες ανεξάρτητες χώρες της περιοχής δυστυχώς και αυτές έχουν διακοπεί. Οι επιχειρήσεις κανονικά θα πρέπει να επιλέγουν τις αγορές τις οποίες θα διαθέτουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανατολικό μας αυτό εταίρο, τη Μολδαβία, όχι μόνο για την εφαρμογή ε, των κανόνων της Συμφωνίας Σύνδεσης αλλά να δούμε και τι άλλες ανάγκες μπορεί να καλύψει αυτή η χώρα. Και γι' αυτό έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις σε προσωρινό επίπεδο που είναι θα έλεγα μία προσωρινή ενδιάμεση μορφή ανακούφισης τομέα των επιτραπέζιων μήλων και των δαμάσκηνων και των επιτραπέζιων σταφυλιών. Αυτά τα οποία προτείνουμε σήμερα είναι προσωρινά μέτρα και θα κρατήσουν για ένα χρόνο. Η πρόταση θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Αύγουστο όταν τέθηκαν οι πρώτοι περιορισμοί ε, στα εξαγωγικά προϊόντα. Ε, τα προϊόντα που εισάγονται δεν θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή αγορά και αυτό διευκρινίστηκε στην πρόταση. Υπάρχουν ανησυχίες βέβαια για τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της ρύθμισης για τους δικούς μας παραγωγούς. Είμαι όμως βέβαιος ότι μπορούμε να στηρίξουμε και να δείξουμε αλληλεγγύη χωρίς ε, εσωτερικές συνέπειες. Οι εισαγωγές ε, μήλων στην Μολδαβία ε, εξαγωγών θα είναι το 0,8%. 1,4% τα δαμάσκηνα και 1,1% τα επιτραπέζια στα φύλλα. Ε, οι μολδαβικές εξαγωγές. Αυτό λοιπόν δεν είναι εμπόδιο για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτή τη χώρα. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ίντε όπως επίσης και τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κανονικά ο κύριος Λαουρένσιο Ρέμπεκα θα το λόγο για ένα λεπτό από την Επιτροπή Γεωργίας αλλά απουσιάζει. Οπότε και θα δώσω μέσα το λόγο στον κύριο Γιούλιο Βίνκλερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Thank you, Chair, uh, Commission. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ΕΛΚ στηρίζει ανεπιφύλακτα τις προτάσεις και νομίζω είναι σημαντικό για άλλη μια φορά να δείξουμε ότι ε, θέλουμε να στηρίξουμε ε, τις γειτονικέ χώρες. Αυτή η έκθεση ε, παρουσιάζει νέα μέτρα για να αντιμετωπιστούν αθέμητες εμπορικές πρακτικές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πέρυσι εγώ ήμουνα εισηγητής της Μολδαβίας όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την πλήρη απελευθέρωση των εισαγωγών κρασιού από τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ε, στυλίτευσε την απαγόρευση αυτών ε, στη Ρωσία. Αυτά που λέμε τώρα είναι το συμπλήρωμα του Περσινού που θέλαμε να ανοίξουμε την αγορά για τα προϊόντα της Μολδαβίας. Συμφωνώ απόλυτα το Κοινοβούλιο να δεχθεί το σχέδιο της έκθεσης χωρίς τροπολογίες αύριο να ψηφίσουμε και μέχρι το τέλος του έτους να δημοσιευτεί η απόφασή μας έτσι ώστε οι εταίροι μας από τη Μολδαβία να επωφεληθούν το συντομότερο δυνατόν. Και κλείνοντας ε, πρόεδρε, ελπίζω ε, στο, να συνεχίσει η ε, Μολδαβία τις προσπάθειές της για σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για την προσέγγιση που υπάρχει με τη Μολδαβία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μάρτινς, David Μάρτινς για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με συγχαρητήρια προς τον κύριο Μόισα. Εξαιρετικός ο εισηγητής και νομίζω ότι είναι η πρώτη του έκθεση παρθενική και τον κύριο Βίνκλερ βεβαίω ω και ο Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο δείχνει ότι ταχεία είναι η αντίδρασή του στι συνθήκε αυτές και είναι καλή συμφωνία που επιτύχαμε. Βοηθήσαμε τη Μολδαβία ε, με τη γεωργική υποστήριξη για τα τρία φρούτα που ακούσατε και ταυτόχρονα αυτό δεν βλάπτει καθόλου ή πάρα πολύ λίγο την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Δηλαδή είναι αμοιβαίω επωφελή αυτή η συμφωνία. Έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τη Μολδαβία για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία απέναντι στην ρωσική επίθεση ε, και την, ε, το εμπάργο αυτό που τους έχει επιβάλει εμείς θα συσφίξουμε τους εμπορικούς μας δεσμούς και θα ενθαρρύνουμε την πολιτική σταθερότητα στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτιν. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Γιασκίεβιτ, Γιασκίεβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, πολύ ε, ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση ε, που κάνουμε για την συμφωνία με τη Μολδαβία. Οι περισσότεροι από εμάς ε, χαιρετήσαμε την ένταξη της Μολδαβίας στις δημοκρατικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι η δημοκρατία της Μολδαβίας εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει στρατιωτική παρουσία των Ρώσων στο έδαφος της και ασκεί πιέσει η Ρωσία και κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε η κυβέρνηση της Μολδαβίας να είναι στα χέρια της και να ε, υπάρχουν ε, ε, αποσχιστικές τάσεις. Ένα άλλο τώρα μέσο πολιτικού εκβιασμού που βρήκε η Ρωσία είναι το εμπάργο στα φρούτα και από την Πολωνία και θα απορροκυπευτικά, όχι μόνο από τη Μολδαβία. Χρειάζεται βοήθεια η Μολδαβία για να μην εξολοθρευτεί η οικονομία της και την αφήσουμε έρμεως στα χέρια του Πούτιν. Πρέπει να τη φέρουμε κοντά μας. Γι' αυτό ο εμπορικός αυτός αποκλεισμός δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Μολδαβία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις να εγκριθούν. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γινόμαστε μάρτυρες μια κατάστασης που πρέπει να τίνουμε μια χείρα βοηθείας προς τους Μολδαβούς αν δεν θέλουμε η Μολδαβία να ε, καταλήξει η Ουκρανία. Πρέπει να τη βοηθήσουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ε, περιμένω συγγνώμη να τελειώσει η διερμηνία. Επόμενο ο κύριο Οστρεβίτσιου από του Φιλελευθέρου. Για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς πριν από ένα μήνα το Κοινοβούλιο υπερψήφισε την Συμφωνία Σύνδεσης με τη Μολδαβία. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι ξεκινώντας την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας, στόχος μας είναι η χώρα αυτή και το σύνολο της περιοχής να καταστεί περισσότερο σταθερό και να ε, απολαμβάνει ευημερία. Όμως αυτό δεν αρέσει στο μεγάλο αδελφό ε, στην ανατολική πλευρά που αποφάσισε να επιβάλλει εμπάργκο τα γεωργικά προϊόντα της Μολδαβίας. Αυτό βέβαια είναι παραβίαση των εμπορικών υποχρώσεων της, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και αυτό βλάπτει όχι μόνο τους Μολδαβούς αλλά και τους Ρώσους. Σήμερα λοιπόν η απόφασή μας είναι κατ' ουσίαν άλλη μία πράξη αλληλεγγύης με τους Μολδαβούς. Πρώτα απ' όλα, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτούς τις 250.000 ανθρώπους που ζουν από τα οποροκυπευτικά. Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η Γεωργία ε, αντικατοπτρίζει περίπου το 40% της, γεωργίας, ε, της οικονομίας της Μολδαβίας. Έτσι λοιπόν, πολύ αναφέρθηκαν στις πρόσφατες εκλογές. Ε, νομίζω ότι κάνουμε το σωστό βήμα από πολιτικό, οικονομικό και άλλα επίπεδα και σεβόμεθα και την ανθρωπιστική διάσταση του προβλήματος. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε ε, για την εισρωή ε, επιτραπέζιων σταφυλιών, δαμάσκινων και μήλων στι ευρωπαϊκές Αγορέ. Είναι νοστιμότατα και πολύ καλά και για το στομάχι μας. Μπράβο, μπράβο λέει η Πρόεδρος, πολύ ωραία. Επόμενο τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριο Σόλτ, εκ μέρους της ε, ΓΚΟΕ. Πρόεδρο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο μολδαβικός λαός ε, αντιμετωπίζει ε, μια μεγάλη πρόκληση και οικονομική και εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Πώς μπορεί να έχει η κοινωνική ε, προοπτική της χώρας ε, απέναντι σε μια μάχη για την εξουσία των μεγάλων δυνάμεων που συγκρούονται εκεί. Η δική μου ομάδα ε, δεν αντιτίθεται ε, με τις εισαγωγές, αλλά χρειάζονται περισσότερα. Πού είναι οι επενδύσεις, πού είναι οι υποδομές, ε, χωρίς να απογοητεύσουμε τον κόσμο. Ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε σχεδιασμό για την ενίσχυση της μολδαβικής οικονομίας. Πού είναι οι νέες καλές θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ανάγκες και υποχρεώσεις μας. Με τη Ρωσία θέλουμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε στο μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να δημιουργήσει και τις ε, προϋποθέσεις για να μπορέσει η Μολδαβία να αξιοποιεί τον πληθυσμό της. Ε, και έχει έρθει και ο χειμώνα πια. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Ο κύριος Σόλτες από τους Πρασίνους παρακαλώ ευχαριστώ πολύ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. θέλω να υποστηρίξω και εγώ την πρόταση αυτή. για τις εμπορικές προτιμήσεις με την, προς τη δημοκρατία της Μολδαβίας έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση το, η Συμφωνία Σύνδεσης που συνεπάγεται στενότερη συνεργασία και πιστεύω ότι με τη συμφωνία αυτή μπορεί και η δημοκρατία της Μολδαβίας να ε, βελτιώσει την πρόσβαση της ευρωπαϊκής αγοράς και να μειώσει την εξάρτηση της από τη ρωσική αγορά. Και αυτό νομίζω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει και στην προσαρμογή της νομοθεσίας ε, στην ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν μόνο θετικές συνέπειες. Η Μολδαβία θα βρεθεί σε μια δύσκολη θέση σε σχέση με την απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών προς τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν θα σημάνει σημαντική οικονομική πίεση και θα φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε την ευθύνη να στηρίξει και σε επίπεδο τεχνοκρατικό αλλά και σε ε, τεχνογνωσίας αλλά και σε επίπεδο οικονομικό τη Μολδαβία. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους, ε, ως μια εγγεγραμμένος ο κύριος Σάνεμανς. Ευχαριστώ. Εγώ συμπαθώ τον ε, μολδαβικό λαό, αλλά σας παρακαλώ συνάδελφοι σταματήστε πια. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλε αυτέ οι φέρπουσε αποφάσει προ την κατεύθυνση αυτή. Τώρα έχουμε και τη Μολδαβία. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Οι ψηφοφόροι δεν συμφωνούν και σίγουρα δεν συμφωνούν οι αγρότε σα. Εσείς συνεχίζετε. Θα πρέπει να μην γελιέστε. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Πού είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης. Είναι σκέτη καταστροφή αυτά που ειναι το οραμα τη ευρωπαικη ενωση ποια ειναι τα ανατολικα συνορα τη ενωση ειναι σκετη καταστροφη αυτα που κανετε Και οικονομικά και από πλευρά ασφαλεία μετανάστευση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε και τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Καλή είναι η συνεργασία με αυτό τη σχεδόν αναπτυσσόμενη χώρα, αλλά ε, με ανεξαρτησία και να σταματήσει από την πίσω πόρτα ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστιαν Νταν Πρέντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης διότι ε, προβλέπονται τρεις ε, φορολογικές απαλλαγές για τα οποροκυπευτικά και έτσι δείχνουμε πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει μια χώρα η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις ρωσικές κυρώσεις και αυτό έγινε κατά της ε, Μολδαβίας ιδιαίτερα. Πρόκειται για μια χώρα η οποία ζει από αυτές τις ε, δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλλιέργεια κυπευτικών. Αυτό δείχνει έλλειψη ανθρωπιάς Δεν μπορούμε να στιγματίζουμε τους ε, φτωχούς οι οποίοι έχουν πληγεί από τους Ρώσους. Αν και εμείς τους πλήξουμε επιπροσθέτως, ε, τότε δεν ε, δείχνουμε ενσυναίσθηση για το τι συμβαίνει στο λαό αυτό. Θα ήθελα να πω ότι οι εκλογές στη Μολδαβία επιβεβαίωσαν την θέληση των πολιτών σε αυτή τη χώρα να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή οδό παρά το γεγονός ότι η Ρωσία χρηματοδότησε και πολιτικά κόμματα κατά ε, της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πιτσούλα έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι εμπορικέ προτιμήσεις είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για τους φιλοευρωπαϊστές εκείνους της Μολδαβίας που μπορούν να προχωρήσουν σε έναν ευθύ δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Μπορεί το θέμα των ποσοστώσεων να αποτελεί μια μικρή οικονομική παραχώρηση προς τη Μολδαβία, αλλά και πολύ σαφές πολιτικό μήνυμα για την ίδια τη χώρα αλλά και τη Ρωσία, για να ξέρει ποιοι είναι ή εταίροι και ποιοι στέκονται δίπλα στη Μολδαβία. 40% του προπολογισμού τη Μολδαβία προέρχεται από τι γεωργικές διαστηριότητε. Και εκεί απασχολείται πολύ μεγάλο ποστό του εργατικού δυναμικού. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι το οικονομικό πλήγμα του εμπάργκο μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειε. Τα ανατολικά σύνορα τη Ένωση παίρνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι πρόσφατες εκλογές δείχνουν ότι η Μολδαβία τάσεται αποφασιστικά υπέρ τη Ευρώπη. Είναι μια μικρή φιλοευρωπαϊκή χώρα και αυτό αποτελεί μια σαφή βάση για το μέλλον μας. Έχει, επιλέξει το δρόμο της Μολδαβία και πρέπει να τη στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πιτσούλα. Ο κύριος Ουιαζδόφσκι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι και αποτελεσματική και θετική. Θα ήθελα να πω όμως στην περίπτωση της Μολδαβίας θα πρέπει να πούμε σαφώς ότι ήμασταν συνεπείς στη δραστηριότητά μας και ήμασταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Δώσαμε μία ευκαιρία στο κράτος αυτό να συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Χαρήκαμε ιδιαίτερα με τη Συμφωνία Σύνδεσης με τη Μολδαβία και σήμερα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το μέσο ελευθέρου εμπορίου είναι πολύ θετικό και έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε τους, αυτούς που τάσσονται υπέρ της Ευρώπης στη Μολδαβία. Επίσης αποτελεί μια πολύ καλή απάντηση στο ρωσικό εμπάργο. Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου με τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία που έδωσαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Με την ευρύ αυτή συμμαχία που τάσεται υπέρ της Ευρώπης. και που καταδικάζουν το, τους ευρωπαϊκούς εγωισμούς. Θα πρέπει να είμαστε ελέγγυοι. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε. Καταρχήν θα στηρίξω την προτυπώμενη τροπολογία προς τον κανονισμό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη Γεωργία η Μολδαβία και αν δώσουμε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο γεωργικό της κόσμο θα στηρίξουμε την οικονομία της. Αυτό όμως που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι πως τα πλεονεκτήματα τα οποία θα δρέψει η Μολδαβία θα φτάσουν ε, και στους ε, καλλιεργητές ε, δαμάσκηνου, μήλων και επιτραπέζιων σταφυλιών. Ξέρετε πως εδώ και έξι μήνες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη κρίση και έχουν χρειαστεί να βρουν καινούργιες αγορές. Στην πραγματικότητα όμως και στην πράξη δεν έχουμε καταφέρει πολλά. Για τα δαμάσκηνα και τα επιτραπέζια στα φύλλα πρέπει να σας πω πως το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η κατάσταση όμως στην αγορά του μήλου είναι πραγματικά δύσκολη. Ευχαριστώ. Ο Αγαπητοί συνάδελφοι, αν υποφέρει αυτή τη στιγμή σήμερα η οικονομικά η Μολδαβία που κανείς δεν το αρνείται, είναι λόγω των επιπτώσεων ε, της απόρριψης της ίδιας της ταυτότητάς της. Το ίδιο πρόβλημα το οποίο έπεσε θύμα η Ουκρανία. Ε, πιέζοντας τη Μολδαβία να διαλέξει στρατόπεδο, δύση, Ευρώπη, δηλαδή προς το στρατόπεδο του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, όπως κάναμε και για την Ουκρανία. Αυτό που κάναμε ήταν να δώσουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, με αποτέλεσμα να θίγεται η τόσο έφραστη αυτή σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο κοινωνία. Αυτές οι μονομερείς, ε, ε, οι μονομερείς ε, κυρώσεις προς τη Ρωσία προκάλεσαν τις αντιδράσεις της Ρωσίας και δεν υπήρχε λόγος ε, για να γίνουν. Τώρα χρειάζεται να δώσουμε κάποιες νέες δυνατότητες στη Μολδαβία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Και αυτή η νέα διάσπαση της Ευρώπης, ε, ο νέος ψυχρός πόλεμος, αυτή η υποστήριξη του ΝΑΤΟ τελικά είναι αντιευρωπαϊκή. Ο κύριος Γκάλερ είναι επόμενος ε, ομιλητής για ένα λεπτό. Μιλά η Μόσχα. Η Μόσχα. Νομίζω αυτά μας είπε ο συνάδελφος κύριος Σαουφράουτζεν. Το θέμα είναι πρέπει να δούμε αν ε, μπορούμε να υποχρεώνουμε κανέναν, αν μπορεί να υπάρχει ο εξαναγκασμός. Ο εξαναγκασμός ε, θα πρέπει να στρέφεται προς τη Μόσχα, τη Ρωσία, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι άλλοι έρχονται εθελοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, Γιατί εμείς υποστηρίζουμε τις ιδέες του κράτους δικαίου και της ευημερίας και όχι τις επεπαλαιωμένες δομές της Σοβιετικής Ένωσης. Εμείς με τις αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις αντιδρούμε σωστά στις πιέσεις της Μόσχας με την πολιτική επιλογή των, εμπορικών, των της αγωγών των γεωργικών προϊόντων που έχει επιβάλει εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια γενική πολιτική εις βάρος της Μολδοβίας. Εμείς θέλουμε να προβάλλουμε και τα μεγαλύτερα ζητήματα. Να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που θα μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουν ταχύτατα τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου και την διαχείριση του κράτους. Αυτά άλλωστε είναι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού προτύπου σε όλους του τομείς της ζωής. Εμείς ξέρουμε ότι το δικό μας μοντέλο είναι αυτό το οποίο δίνει, δείχνει το δρόμο προς το μέλλον στον άνθρωπο και είναι η σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλερ. Η κυρία Κανιέτε. Και πριν σας δώσω το λόγο κυρία Κανιέτε, θέλω να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά για την ομιλία σας. Γιατί είστε η μόνη γυναίκα που λαμβάνει το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Από τους βουλευτές, από τους βουλευτές κυρία Επίτροπε. Um, ευχαριστώ πολύ. Είμαι περήφανη. Είμαι περήφανη λοιπόν που είμαι γυναίκα. Και θα συνεχίσω στα λετωνικά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο και να σας πω πως το σύστημα αυτό προς τη Μολδαβία αυτή η προσφορά δεν έχει μόνο οικονομική σημασία αλλά έχει και πολιτική σημασία δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πως έχει τη δυνατότητα να δράσει υπέρ της δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Και αυτές οι προτιμήσεις θα προσφέρουν άμεση ανακούφιση στη μολδαβική οικονομία χωρίς να επηρεάσουν καθόλου την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιδράσει στις προσπάθειες του Πούτιν να τιμωρήσει τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία προτιμούν την οδό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πριν από μερικές εβδομάδες κοινοβουλευτικές εκλογές στην ε, Μολδαβία έδωσαν ένα ξεκάθαρο νικητή τις προευρωπαϊκές δυνάμεις και φανταζόμαστε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να υπάρξει ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση στην Μολδαβία και η Μολδαβία να είναι πια ένα πετυχημένο παράδειγμα. Είναι ένα πολιτικό σήμα λοιπόν, μήνυμα που στέλνουμε στην Μολδαβία που δεν μπορεί βέβαια να υποκαταστήσει αυτές τις προοπτικές μιας ξεκάθαρης δυνατότητας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς πολλά κρατημέλη και πολλοί ευρωβουλευτές δεν είναι έτοιμοι ακόμα για να προσφέρουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε το Ευχαριστώ κύριε Κανιέτε. Ο κύριος Λαντσπέρκης για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε τόσο αργά. Εδώ και μερικές εβδομάδες έγινε λόγος για μία συμφωνία ε, κοινού εμπορίου με τη Ρωσία που αρχίζει από το Βλαδιβοστόκ και τελειώνει στη Λισαβόνα. Δεν πρέπει να ε, ξεχνάμε τη συμφωνία που άρχισε από το Βανκούβερ και τελειώνει στο Κισινάου ή περνάει μέσα από την ε, τυφλίδα. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη διακίνηση των αγαθών. Μετά τις εκλογές στην Ουκρανία και τη Μολδαβία βλέπουμε ότι οι δύο χώρες αυτές θέλουν να ακολουθήσουν τη δημοκρατική οδό και ακολουθούν μια φιλοευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ κύριος Στήρ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω τη διαδικασία διαδικασία εντατικοποίησης πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας. Βεβαίως υπογραφή της, σύμβασης, ε, της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης τον Ιούνιο ήταν πολύ θετική γιατί εντατικοποιούνται αυτές οι προσπάθειες συνεργασίας, αλλά δεν θα πρέπει να μην λάβουμε υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις και τη στάση της Ρωσίας. Η Μολδαβία ακολούθησε τη δική της οδό, κάτι το οποίο θεωρήθηκε απαράδεκτο από τη Ρωσία που τη θεωρεί δορυφόρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και αυτό αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τον αποκλεισμό τους. Αυτό έπληξε αρνητικά την οικονομία διότι ο γεωργικός τομέας είναι πολύ σημαντικός. Το 10% του εργατικού δυναμικού ασχολείται με τα οποροκυπευτικά. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα δαμάσκηνα, τα μήλα και τα επιτραπέζια σταφύλια στο κανονισμό ελευθέρου εμπορίου γιατί έτσι θα βοηθήσουμε τους μικρομεσαίους παραγωγούς και θα αποστείλουμε και ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία. Θα δείξουμε δηλαδή αλληλεγγύη με τη Μολδαβία. Ευχαριστώ κύριε Στήρ. Ένα μισή λεπτό κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συχνά μου λέμε ότι οι πολιτικοί σε όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ψυχή ή καρδιά. Αλλά όταν βλέπουμε αυτές τις προτάσεις νομίζω ότι φαίνεται και πως έχουμε και καρδιά και ψυχή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δουλέψουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα. Εφαρμόζουμε μέτρα απαραίτητα αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα για τους φτωχότερους κατοίκους της Μολδαβίας, για τους γεωργούς που υποφέρουν διότι οι πολιτικές που επιβάλλονται υπό την επιρροή του Βλαντιμίρ ε, Πούτιν ε, τους ταλαιπωρούν. Όπως υπόθηκε και από την Επιτροπή πρέπει να πληχθούν νέε δυνατότητες για τις αγορές. Αυτό όμως δεν γίνεται μέσα σε μια νύχτα. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσει τη βοήθεια προς τους γείτονές μας και πρέπει με τον τρόπο αυτό να αποδείξουμε πως έχουμε καρδιά, πως έχουμε ψυχή. Ακόμα περισσότερο. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε και χωρίς να επιβαρυνθούν δικοί μας Γιώργη. Γιατί όπως είπε και η Επίτροπος, πρόκειται για, το, για ποσοστό μικρότερο του 1% σε σχέση με την αξία των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πολύ καλή η πρόταση. Και δείχνει όπου όπως λέμε στα αγγλικά ότι στην ανάγκη φαίνεται ο φίλος. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δείξουμε στη Μολδαβία, ότι όταν μας έχει ανάγκη είμαστε φίλοι της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Τελευταίος ομιλητής του καταλογό μου, ο κύριος Αντρέι Τζιπ, για 1,5 λεπτό. Το σύστημα αυτών των προτιμήσεων είναι ένα εργαλείο το οποίο το προβλέπει και η ίδια η πολιτική γειτονίας. Και σε αυτό το εργαλείο ε, προσφεύγουμε κάθε φορά που δεν έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους εταίρους μας παρά μόνο ε, τροποποιώντας ε, το σύστημα αυτό των προτιμήσεων έτσι ώστε τα πλεονάσματα σε δικά τους εμπορεύματα τα οποία θα πήγαιναν σε ρωσική αγορά να μπορούν οι Μολδαβοί φίλοι να πουλήσουν σε ευρωπαϊκές αγορές. Η Μόσχα αντέδρασε με πολύ στεναρό τρόπο και ακούσαμε βέβαια το τι συμβαίνει και πώς αντιμετωπίζουν τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Μολδαβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή δηλαδή η ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών όπως επίσης και η απελευθέρωση κάποιων ε, ε, ε, ε, η απελευθέρωση κάποιων εξαγωγών δημιούργησαν προβλήματα. Ελπίζουμε πως με τις νέες αυτές προτιμήσεις θα επιτρέψουμε να σταθεί κάπως τα πόδια το κλάδο της γεωργίας στη Μολδαβία, στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού της χώρας. 13 Σεπτεμβρίου έγιναν εκλογές βουλευτικές. Εγώ Πήγα στη χώρα λίγο πριν τις εκλογές και πολλοί κόσμοι μου είπε πως ανησυχεί λόγω του εμπάργου που τους έχει επιβάλει η Ρωσία. Πιστεύω πως η ταχεία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα κομμάτια της μολδαβικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα δεν βλέπω ούτε άντρα ούτε γυναίκα βουλευτή να ζητάει το λόγο με τη δικασία Καριστιά. Παρακαλώ την κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριε και κύριοι βουλευτέ, νομίζω ότι η απόψινη συζήτηση επιδεικνύει σαφή και ισχυρή έλεγγυη. Ένα πολύ καλό δείγμα, Μόλι πριν από τα Χριστούγεννα. Όπω είπαν όλοι οι ομιλητέ, σχεδόν. Είναι προφανέ ότι δεν επηρεάζει τη δική μα αγορά. Πρόκειται για 0,1% του ε, εμπορίου. Είναι πολύ σημαντικό όμω για τη Μολδαβία οικονομικά αλλά και πολιτικά. Η αλληλεγγύη λοιπόν αποδεικνύεται πως δεν είναι απλώς λέξη καινή για μας, αλλά ένας τρόπος να στηρίξουμε πραγματικά τους γειτονές προς Ανατολάς. Ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία στην έγκριση από το Κοινοβούλιο και έτσι θα δείξουμε ότι οι χώρες που επιλέγουν το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης και τις ευρωπαϊκές αξίες ε, ε, έχουν υποστηρικτεί και στήριγμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν φίλου σε δύσκολε εποχέ. Όχι μόνο η Μολδαβία, αλλά όλε οι χώρε. Και θα συνεχίσουμε να τη βοηθούμε τη Μολδαβία και στο μέλλον και θα παρακολουθούμε με προσοχή την ε, λειτουργία της συμφωνίας, η οποία θα εγκριθεί ελπίζουμε αύριο. Ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και την Επιτροπή για τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Για άλλη μια φορά τώρα ο κύριος Μωυσά θα πάρει το λόγο, ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο η οποία εργάστηκε τάχιστα επί του θέματος αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεισέφεραν απόψε στη συζήτηση. Βλέπω ότι υπάρχει κοινή λογική ε, στην πλειοψηφία των αντιδράσεων και Θεωρώ ότι η μόχλευση είναι μία λέξη του σειρμού. Νομίζω λοιπόν ότι με μία προσπάθεια θα φτάσουμε σε έναν λόγο 1 προς 15 και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τους Μολδαβούς. Ως προς τα σχόλια που αναφέρθηκαν, κύριε Σόλτς, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, Συμφωνία Γενικευμένων Προτιμήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει προστιθέμενη αξία προς τους Μολδαβούς. Θεωρώ ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια και των ευεργετημάτων της ενίας αγοράς σε σχέση με τη διεύρυνση αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ε, το δικαίωμα άρνηση κυρίας, γι' αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε ένα κανονισμό παρά μόνο σε ορισμένα προϊόντα. Μιλάμε για τα δαμάσκηνα και τα μήλα. Βεβαίως η Μολδαβία θέλει να προσχωρήσει στην Ευρώπη και οι, πολιτικοί παίκτες μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την δημοκρατική διαδικασία. Ο κύριος Σαφχάουζερ. Ε, στην ουσία τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι το θύμα είναι υπεύθυνο του βιασμού. Μιλάμε για άρνηση της ε, μολδαβικής ταυτότητας, μα αυτό είναι παράλογο. Κανένας δεν υποχρεώνεται ε, Μολδαβία να προβεί σε μια επιλογή. Επιλέγει αυτό που επιθυμεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα χώρα αύριο.